Good morning Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάει η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα αναβάλλεται, η κοινή συνεδρίαση με την ΕΚΟΝ. Οπότε τώρα το πρώτο θέμα είναι η έγκριση ημερήσιας ε, διάταξης. Ε, ε, σας στείλαμε χθες ε, την ημερήσια διάταξη, αναθεωρημένη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνεται. Δεν βλέπω κάποια αντίρρηση. Το επόμενο θέμα ανακοινώσει του Προέδρου. Το πρώτο θέμα είναι η ακύρωση της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου. Η συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται, ακυρώνεται μάλλον. Είχαμε... Η δε συνεδρία στις 27 Φεβρουαρίου θα λάβει χώρα κανονικά. Θα σας στείλουμε εν καιρό την ημερήσια διάταξη η διερμηνία. Ε, υπάρχει σε 20 γλώσσες, δηλαδή δεν υπάρχει στις βαλτικές γλώσσες ε, και την ε, γοεδαλική. Η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο και βεβαίως ε, αυτό γίνεται ήδη και μέσω της εφαρμογής e-meeting. Το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε ή μάλλον για το οποίο θα σας ενημερώσω αφορά τις ε, διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Έχουμε δύο θέματα στο Συμβούλιο. Το ένα αφορά τους επίμονους οργανικούς ρήπους στις 19 ε, Φεβρουαρίου είχαμε τον τρίτο και τελευταίο τριμερή διάλογο. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κατάληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία για ολόκληρο το νομοθετικό κείμενο. Αφορούσε δε, το παράδειγμα 4 και τα όρια συγκέντρωσης ουσιών και τα μέσα τροποποίησης, όπου η πρόταση της Κομισιόν επιβεβαιώθηκε από την εντολή του Κοινοβουλίου και τα όρια αυτά παρουσιάζονται στα παραρτήματα και τις πράξεις κατεξιοδότηση αφενός και αφετέρου έχουμε την εντολή του Συμβουλίου και την διαγραφή των ορίων συγκέντρωσης από τα παραρτήματα και την ε, εφαρμογή τους μέσω εφαρμοστικών πράξεων. Είχαμε λοιπόν την τακτική ε, νομοθετική διαδικασία την οποία εμείς προτείναμε. Η Κορεπέρ ε, θα το συζητήσει την Παρασκευή, το συζήτησε 22 Φεβρουαρίου, ενώ εμείς, ε, όχι θα το συζητήσει 22 Φεβρουαρίου, ενώ εμείς θα το ψηφίσουμε στις 29 Φεβρουαρίου. Το άλλο θέμα είναι οι εκπομπές διοξείδου του άνθρακα από βαρέα οχήματα ο τέταρτος και τελευταίος ε, διάλογος για το θέμα αυτό. Εκεί πέρα Συμβουλή και Κοινοβούλιο κατάφεραν να συμφωνήσουν. Η τελική συμφωνία, η οποία επιτευχθεί νωρίς το πρωί, είχε τα εξή στοιχεία. Για το EMS, το Συμβούλιο συμφώνησε να προσθεθεί το EMS στο άρθρο 13 ναι, όσον αφορά το ζήτημα που αναφέρει το εκτιμώ 34. Το ύψος των εισφορών για την υπέρβαση των εκπομπών, το Κοινοβούλιο δέχτηκε 4.500 ευρώ αναγραμμάριο διοξιδίου του άνθρακα χιλιόμετρο για την περίοδο 2000 25-2045. Για το 2025 δεχτήκαμε μία μείωση 15% και 30% μείωση από το 2030 ε, κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί στην αξιολόγηση του 2022 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων. Οι αριθμοί αυτοί συμφωνήθηκαν με αντάλλαγμα ακριβώς ενός συστήματος συγκριτική αξιολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων με ένα 2% από το 2025. Τέλος, συμφωνήσαμε το να μην βασιζόμαστε στα ονομαστικά νούμερα για τις ε, εκπομπές ε, των ηλεκτρικών οχημάτων. και σκοπεύουμε όλα αυτά να πάνε στην Ολομέλεια την 2η του Απριλίου. Το επόμενο θέμα είναι η κοινή συζήτηση τριών διαφορετικών αντιρρήσεων για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πρώτα απ' όλα λοιπόν οι συνεισηγητές θα έχουν την ευκαιρία να παρέμβουν Πρώτα απ' όλα, όπως συμφωνήσαμε, η κυρία Ελεονόρα Εύη θα λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για μια φορά ακόμα τις αντιρρήσεις μας για το γενετικό τροποποιημένο αραβόστο που θέλει να βάλει σε εμπορία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν εγκριθεί σήμερα και το Μάρτιο, θα φτάσουμε στις 34 αντιρρήσεις σε αυτή τη θητεία για την Επιτροπή μας συνολικά, μαζί με τις υπόλοιπε τρει, που είναι το υψηλότερο ρεκόρ που είχαμε. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί, παρόλε τις αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει αυτά τα γενετικά τροποποιημένα. Εμείς έχουμε εκλεγεί από τον Ευρωπαϊκό ελληνικό και συνέχεια λέμε όχι. Και δεν βρίσκεται ποτέ η ειδική πλειοψηφία που να είναι υπέρ. Παρ' αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να τα περάσει και υπάρχουν και διαδικαστικά προβλήματα αλλά και ε, προβλήματα με τις εξασφαλίσεις που δίνονται για αυτούς τους γενετικώς ε, για αυτά τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα ε, στους Ευρωπαίους καταναλωτές ε, ότι είναι ασφαλή. Καταρχήν, οι τρει αυτοί ε, ε, γενετικώς τροποποιημένοι αραβόστοι ε, ε, παρουσιάζουν ε, προβλήματα με παρουσία γλυφοσάτη που είναι καρκινογόνο ουσία και δεν έχει γίνει η κατάλληλη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιολογήσει κατά πόσο δικαιολογείται η έγκριση ή η απόσυρση τη έγκριση. Για τα γλυφοσυνάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σα πω ότι πλέον δεν επιτρέπεται γιατί είναι τοξικά για την αναπαραγωγή και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να δίνει έγκριση για τέτοιου είδου φυτά τα οποία έχουν ψεκαστεί ε, σε τρίτε χώρε με γλυφοσυνάτη. Και νομίζω ότι και αυτοί οι τρει γενετικώ τροποποιημένοι αραβόσιτοι ε, θα έχουν ε, ε, ε, ε, ψεκαστεί με γλουφοσυνάτη και θα έχουν πολύ περισσότερα κατάλοιπα για το λόγο αυτό. Πρέπει να σου πω στα κατάλοιπα αυτά και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σε συνδυασμό με το γενετικό τροποποιημένο ραβόστο δεν έχουν ληφθεί υπόψη δεόντως στην συζήτηση για την αξιολόγηση και γι' αυτό έχουμε ζητήσει να δούμε τον την έκθεση ε, αξιολόγησης κινδύνου για όλα τα παραπάνω, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Σε προηγούμενε συζήτησεις που έχουν γίνει για τέτοιου είδου αντιρρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε συχνότητα πω οι Ευρωπαίοι πολίτε είναι ασφαλεί από ε, τις συνέπειες από τέτοιου είδου κατάλοιπα άλλων ζυζανιοκτώνων, γιατί τα ανώτατα όρια γίνονται ε, ε σεβαστά. Αλλά εμεί ξέρουμε πω αυτά τα μέγιστα ε, κατάλοιπα δεν λαμβάνουν υπόψη γεγονό πω μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί πάνω ένα είδο ζυζανιοκτώνου, δύο ή και παραπάνω, και είδαμε πω για κάποια εντομοκτένα, για παράδειγμα για τη γλυφοσάτη, ο ορισμό του, ε, του μέγιστου ε, ε, επίπεδου ήταν αρκετά χαμηλότερο από τον αριθμό παραδειγμάτων που θα έπρεπε να έχουν αναλυθεί για να μπορούμε να έχουμε κάποια επιστημονικά πραγματικά ασφαλή δεδομένα. Για την περίοδο 2020-2021 και τις εγκρίσεις που έχουν δεθεί δεν υπάρχει υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να ε, ελέγχουν αν έχουν ε, κατάλοιπα γλυφοσάτης ή γλυφοσινάτης αυτή η εισαγόμενη αραβόσιτη. Για τη βιώσιμη χρήση ε, ζύζανιοκτώνων εμείς ζητήσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνεται περισσότερος έλεγχος για προϊόντα τα οποία έχουν ψεχαστεί με ζυζανιοκτώνα τα οποία απογαρεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα γλυφοσινάτη. Η ερώτηση μου είναι λοιπόν εδώ η Κομισιόν τι θα κάνει και για τη δεύτερη και τρίτη αντίρρηση που έχουμε για τους δύο αυτούς αραβόσιτους με τους κωδικούς που βλέπετε και για τους συνδυασμούς αυτών να σας πω τα εξής. Ανησυχούμε για την καταμειοψηφία ε, γνωμοδότηση του ε, πάνελ, τον Μισελ ε, Γιατί? τέτοιου είδους ε, αποφάσεις κατά μειοψηφία ε, παρουσιάζονται μόνο όταν υπάρχουν σημαντικές αντιρρήσεις. Γιατί προσπαθεί να αποδείξει ο επιστήμονας αυτός πως οι βιοτοξίνες που χρησιμοποιούνται για τις ε, δράσεις τους μπορεί να κάνουν υψηλότερη την αλληλογόνα ε, επίδραση άλλων τροφίμων. Και στην ε, έκθεση αυτή μειοψηφίας αναφέρεται πως η ΕΦΣΑ δεν κάνει τα απαραίτητα, τις απαραίτητες για να εντοπίσει τα κατόφλια αυτά. Επίσης, αυτή η έκθεση καταλήγει ότι δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί ο ρόλο των γεννητικά τροποποιημένων οργανισμών σε, ε, στην αύξηση του ε, αλλεργιογόνου κίνδυνου και με τον τρόπο αυτό δεν προστατεύονται απόλυτα οι καταναλωτέ οι οποίοι ενδεχομένω βρίσκονται σε κίνδυνο. Και αυτά τα λέω γιατί υπάρχει πρόβλημα ε, με τον αραβόσιτο που έχει κατάλοιπα τέτοιων ζυζανιοκτώνων και που πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν αλληλικέ αντιδράσει καταναλωτέ. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί η Κομισιόν θέλει να επιτρέψει την είσοδο αυτών των προϊόντων. Uh, για τους σοσιαλιστές, κυρία Κάντεμπαχ, ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ομιλώ σήμερα εκ μέρους του κ. Μπαλάς. Ήθελα να ξεκινήσω με ένα γενικό σχόλιο για τις... Ε, αντιρρήσει ε, για τα γενετικώ τροποποιημένα. Όλε οι αντιρρήσει μα έχουν ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Αντιρρήσει που έχουν υποβληθεί από εκπροσώπου έξι πολιτικών ομάδων, ε, σοσιαλιστέ, ε, Γκουε, Άλντε, EFTD. Η πλειοψηφία ε, ψήφισε μια τροπολογία που ζητά να αναθεωρήσει η Κομισιόν την πρότασή της ε, για τοποθέτηση των GMO στην αγορά. Στόχος μας είναι να μην έχουμε γενετικώ τροποποιημένα προϊόντα εγκεκριμένα στην Επιτροπολογία εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει νέα πρόταση ε, για να ληφθεί υπόψη η επίδραση στην Ευρώπη. Είναι θέμα δημοκρατίας. Οι αντιρρήσει αυτέ είναι ένα τρόπο επίση να διασφαλίσουμε ότι οι επιλογέ του Κοινοβουλίου θα γίνουν σεβαστέ. Ε, στο πλαίσιο των θεσμικών του προνομίων. Η αντίρρηση αυτή δεν έχει άλλο σκοπό παρά την εφαρμογή της εφαρμογής της προφύλαξης ε, ε, το σεβασμό τη πλειοψηφία μια αιρετή συνέλευση, διαφάνεια και δημοκρατικέ επιλογέ ώστε να αποκατασταθεί μια Ευρώπη η οποία προστατεύει του πολίτε τη. Εμεί θέλουμε να χρησιμοποιηθούν οι Πιστεύουμε ότι οι άδειε αυτέ θα οδηγήσουν σε κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων, την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και για το περιβάλλον. Σύμφωνα με, όπω και στι προηγούμενε αντιρρήσει, θεωρούμε ότι η Επιτροπή, αναγνωρίζοντα τα σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, όπω εξηγείται στην αιτιολογική ε, ε, σκέψη της πρότασης συνεχίζει να επιτρέπει την κυκλοφορία των ε, γενετικώς τροποποιημένων ουσιών. Δεν έχουν δοθεί γνωμοδοτήσει από καμία επιτροπή ε, και έχουν απορριφθεί οι προτάσεις αυτές από το Κοινοβούλιο. Η τοποθέτηση στην αγορά ε, προϊόντων ε, από γενετικό τροποποιημένο αραβόσιτο λόγω της αντοχής ορισμένων ε, οργανισμών ε, ε, του γραφιά του Αραβόσιτου στο πλαίσιο του DSRNA ενός εντομοκτώνου το οποίο έχει επίδραση ότι προσλαμβάνεται στο έντερο του οργανισμού, στην ύμφη αυτού του γραφιά του αραβόσιτου και διαταράσει τις βιολογικές διαδικασίες, σκοτώνοντας ε, το γραφιά αυτών. Ωστόσο, η ΕΦΣΑ έχει περιορίσει τις, ε, την αξιόλογηση κινδύνου σε πιθανές παράπλευρες ε, επιδράσεις στα φυτά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις στους ανθρώπους, στα ζώα κτηνοτροφίας και στα άλλα ζώα που εκτίθενται σε αυτό μέσω της διατροφικής αλυσίδας. Μια γνωμοδότηση από την Tex 10 ένα ανεξάρτητο οργανισμό, το περιγράφει ως ένα τέλειο παράδειγμα ε, όπου κάνουμε τα στραβά μάτια. Ε, αυτό δεν συνάδει με τις υπάρχουσες ε, νομοθεσίες. Επίσης αυτό έχει αντοχή στο γκλέφοσατ. Το 060244 αφορά την τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων από ε, ενός συγκεκριμένου ε, BT11MIR e 162-1507-GA21 και επιμέρους συνδυασμούς BT11MIR 162-1507-MIR 162-1501-GA21 και MIR 162 και 1507. Δεν έχουν δοθεί για κανένα επιμέρους συνδυασμό δεδομένα. Δεν θεωρήθηκαν απαραίτητα για την αξιολόγηση κίνδυνο, ωστόσο η ΕΦΣΑ δεν ζήτησε πειραματικά δεδομένα για τους τρει επιμέρους συνδυασμού. Η ε, γνωμοδότηση μειοψηφία υιοθετήθηκε από ε, ε, κάποια μέλη και είπαν ότι η αξιολόγηση των ορισμένων ουσιών δεν, έχει γίνει χωρί απαραίτητα δεδομένα, παρέχοντα την ίδια αξιοπιστία για την αξιολόγηση, όπω και για την αξιολόγηση γενετικώ τροποποιημένων ουσιών, για την οποία έχουν δοθεί δεδομένα. Επίση, η γνωμοδότηση μειοψηφία λέει ότι οι μελέτε δείχνουν ότι έχουν παρατηρηθεί παραπλευρέ επιδράσει που μπορούν να επηρεάσουν το νοσοποιητικό σύστημα ε, λόγω έκθεση ορισμένε ε, πρωτενε BT. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες, ε, κάποιες πρωτεΐνες όπως αυτές έχει αποδεχθεί ότι μπορούν να αυξήσουν την αλλεργιογόνο επίδραση άλλων πρωτεϊνών με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή. Σε κάθε περίπτωση η ε, γνωμοδότηση μειοψηφία ε, λέει ότι παρότι δεν έχουν παρατηρηθεί παρατηρήσεις ε, επιδράσεις ε, δεν, είναι δυνατόν, δεν θα ήταν δυνατόν να έχουν ανεχνευτεί με τις τοξικολογικές μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή για την αξιολόγηση ασφάλειας των ε, φυτών, των γενετικών τροποποιημένων φυτών, διότι δεν έχουν συμπεριληφθεί συγκεκριμένες, τα συγκεκριμένα τεστ για αυτό το σκοπό. Λόγω έλλειψη λοιπόν δεδομένων για τους τρεις επιμέρους συνδυασμού, ο κίνδυνος αυξημένη παρουσίας των πρωτεϊνών BT και των πιθανών σωρευτικών επιδράσεων του συνδυασμού του στο ανοσοποιητικό σύστημα, για παράδειγμα με διάφορες ε, επιδράσεις ε, δεν μπορούν να αποκλειστούν. Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε σαφώς ε, κατά πόσο αυξάνουν την αλλεργιογόνο δράση και κατά πόσο προστατεύονται πλήρως οι καταναλωτές. Αυτοί οι τρεις συνδυασμοί, η αντίσταση σε ζυζανιοκτώνα η... και διάφορες επιδράσεις είναι Σημαντικέ για την ενδελεχή αξιολόγηση κινδύνου για τα φυτά αυτά, τα γενετικώ τροποποιημένα. Ωστόσο, τα κατάλοιπα από ψεκασμό με ζυζανιοκτώνα δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο ε, ε, αρμοδιοτήτων της ΕΜΣΑ για αυτούς τους οργανισμούς. Έτσι λοιπόν δεν έχουν αξιολογηθεί αυτού του είδους τα ζυζανιοκτώνα. Παρακαλούμε λοιπόν την Κομισιόν να μην εξου... Ε, αδειοδοτήσει τέτοιου είδου ε, προϊόντα, εκτό αν εκεί γίνει αξιολόγηση από την ΕΦΣΑ βάσει πλήρων δεδομένων που θα έχουν ε, υποβληθεί από τον Ετούντα. Το 06402 ε, το, ο αραβόστος 114 περιλαμβάνει διάφορες τοξίνες πρωτεΐνες που Ζητά ο Πρόεδρος αν μπορεί να ε, ολοκληρώσει η κυρία Ομιλήτρια. Ουσιαστικά ναι, έχουμε, φέρνουμε ένσταση. It was quicker than I expected, <laughs> but thank you very much. <laughs> It's a clear statement. And then um, in the round of the shadow rapporteurs, I give the floor to... Για τους σχέδιους συζητητές ε, δίνω το λόγο στον κύριο Φιέλνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνοψη αυτή. Λοιπόν, να, πάλι τα ίδια. Τα έχουμε πει ξανά και ξανά. Κοιτάξτε, όταν ε, φέρνουμε αυτές τις ανταρρήσεις ε, έχουμε σκοπό να ελέγξουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αν ξεπέρασε η Κομισιόν την εντολή της, βλέπω ότι κανείς ε, δεν έχει ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο είναι εάν η Κομισιόν δεν άκουσε την επιστημονική γνωμοδότηση. εκεί πέρα ε, είναι η κύρια αντίσταση. Η γεγονός είναι ότι ε, ούτε αυτό ισχύει γιατί το πάνελ της ΕΦΣΑ κατέληξε ότι τα λόγω αυτά προϊόντα είναι εξίσου ασφαλή με τα συμβατικά ε, καλαμπόκια όσον αφορά και το περιβάλλον και την υγεία. Έχουμε τη σκληρότερη νομοθεσία στον κόσμο, την σκληρότερη επιστημονική αξιολόγηση στον κόσμο, αλλά αυτό δεν αρκεί, Οπότε βλέπω. Ε, σημειώνω ότι προσπαθείτε εδώ πέρα να πείτε ότι αυτά δημιουργήθηκαν για να είναι ανθεκτικά στην γλυφοσάτη, την οποία ε, συζητάμε, αλλά δεν απαγορεύεται ακόμα στην Ευρώπη. Ξέρω ότι κάποιοι θέλουν να την απαγορεύσουν, είναι δύσκολο να απαγορεύσουμε κάτι επειδή σχετίζεται με κάτι το οποίο δεν είναι απαγορευμένο. Οπότε πάτε στο επίπεδο καταλήπων. Μα υπάρχει και νομοθεσία για τα κατάλοιπα. Και για να γίνει δεκτό οτιδήποτε πρέπει να πληρεί αυτή η νομοθεσία. Εντάξει, μπορεί να σα πειράζει αυτή η νομοθεσία, αλλά να εστιάσουμε τότε σε αυτήν την νομοθεσία περί καταλήπων. Αντί να απαγορεύσουμε κάτι επειδή σχετίζεται κάτι ε, το οποίο σχετίζεται με κάτι άλλο το οποίο δεν είναι απαγορευμένο. Και τα έχω ξαναπεί αυτά. Αλλά ε, θα τα επαναλάβω όσο τα επαναλαμβάνετε κι εσεί. Ε, επαναλαμβάνετε αυτέ τι ε, γελίε αντιρρήσει. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια υποκρισία. Και έχετε αρχίσει να ακούγεστε σαν αυτούς που αρνούνται την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει εδώ πέρα συνένεση επιστημονική, όχι μόνο για την κλιματική αλλαγή, αλλά για το ότι τα γενετικά τροποποιημένα δεν είναι πιο επικίνδυνα από ότι τα συμβατικά προϊόντα. Εδώ, λοιπόν, βρίσκεται μια ε, μειονότα, κάποιους δικούς σας επιστήμονες που λένε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτήν τη συνένεση. Και, και πάλι, δηλαδή το έχω ξανακούσει και αυτό, ε, και στην κλιματική αλλαγή και ακούγεστε πάρα πολύ σαν αυτούς. Λοιπόν, δεν είναι μια εκστρατεία ε, κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, είναι μια εκστρατεία κατά της χάραξης πολιτικής με βάση την επιστήμη. Ε, δυστυχώς ε, σε αυτήν την παροδία συμμετέχει η πλειοψηφία αυτής της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντελά, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Άκουσα να αναφέρεται αρχή της προφύλαξης. Η αρχή της προφύλαξης δεν είναι για να μην κάνουμε κάποια πράγματα, είναι μια αρχή αναλογικότητας όταν υπάρχει κίνδυνο και ανάλογα με το επίπεδο πρέπει να αναλαμβάνετε τα ανάλογα μέτρα. Η αρχή τη προφύλαξη λοιπόν δεν είναι αρχή αδράνεια. Να το καταλάβουμε καλά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στους ε, ε, μεν στους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αλλά και στις συμφωνίες που μας επιβάλλουν ε, ε, στι συμφωνίε που επιτρέπουν να μην μπουν ε, στον χώρο τη ενιαία αγορά οι ουσίε τι οποίε δεν θέλουμε στην Ευρώπη. Εγώ είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένη λόγω τη συζήτηση. Ο συνάδελφο Φιέλνερ είπε ακριβώ αυτά που είχα και εγώ στο νου μου. Σε αυτά ήθελα να αναφερθώ και εγώ. Εάν δεν θέλουμε γενετικώ τροποποιημένε ουσίε στην Ευρώπη, α μην ε, το λέμε με, προσχε... με διάφορους ε, πλάγιους τρόπους, ας μην τα δεχτούμε. Όχι να επιτρέπουμε σε εκατομμύρια προϊόντα τα οποία παράγονται με ουσίες που δεν επιτρέπεται στην Ευρώπη να μπαίνουν στην αγορά μας και να τρέφουν τους πολίτες μας και τα ζώα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, α, όχι, κυρία Γιούσου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συνταχθώ με τους ε, συναδέλφους. Είναι υποκριτικό να απαγορεύουμε εδώ τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Κανείς δεν κατάφερε να αποδείξει πως έχουν οποιαδήποτε επίπτωση αρνητική στην υγεία ή σε τίποτα άλλο. Και πιστεύω πως ε, εδώ θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή του ότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεν θα επιφέρουν μία αυτόματη αντίρρηση. Γιατί αν το κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να θρέψουμε τα κοπάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν θα υπαρκούσαν οι ζωοτροφές. Ευχαριστώ. Darling. κυρία uh, yes, thank you. Um, well, I... Ευχαριστώ. Okay. έχουμε ξανακούσει αυτά που είπε και ο κύριος Φιέλνερ και δεν έχει αλλάξει ε, τίποτα. Εκτός από, και εδώ πέρα συγχαρώ όσους ε, φέρνουν αντίρρηση γιατί γίνονται και κάπως πιο πιστικοί και λένε όλες τις χημικές ουσίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το σκεπτικό τους είναι σωστό. Ε, και μάλιστα ακούγονται κάπως απεγνωσμένοι. Θεωρώ εγώ. Σαφώς έχουμε εδώ πέρα ένα κυνήγι μαγισσών κατά κάποιων προϊόντων και των ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα παρά το ότι έχουν λάβει άδεια για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θα επεσήμενα ότι φράσεις όπως ε, υπήρχαν ερωτήσεις ε, για το καρκινογόνο του πράγματος της γλυφοσάτης Καταλήξαμε όμως και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν ε, συμβαίνει αυτό. Ήταν ξεκάθαρο το συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτρη δεν είναι καρκινογόνος, αλλιώς δεν θα είχε ξαναπάρει άδεια. Ακούσαμε για την ε, γλυφοσανάτη, εντάξει ξέρω πως οι Γάλλοι την έχουν απαγορεύσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι στην ίδια θέση και δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία ότι οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα καθιονδήποτε τρόπο ε, εμπλέκεται σε οποιαδήποτε καρκινογένεση ε, μέσω ε, ακριβώ αυτών των τροποποιημένων γενετικά προϊόντων. Δηλαδή επειδή ακριβώς ε, μπορούν να ψεκαστούν, δεν σημαίνει ότι ψεκάζει κιόλα και δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο, αλλιώς δεν θα είχαν πέρασει το πολύ αυστηρό ευρωπαϊκό σύστημα έγκρισης. Και πάλι λοιπόν ε, έχουμε κάποιες αρχές, τι οποίες έχουμε κάνει σαλάτα. Και εδώ πέρα να πω ε, στον κύριο Τέλα ότι η αρχή αυτή της προφύλαξης υπάρχει στις συνθήκες ε, όταν δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία. Όχι όταν κάποιο προσωπικά ανησυχεί και λέει Αχ, όχι, τι είναι αυτό το πράγμα. Όταν δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία και δεν υπάρχουν προϊόντα ε, που να έχουν υποστεί περισσότερου επιστημονικού ελέγχου και ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα προϊόντα αυτά. Οπότε να συνεχίσουμε ε, να λέμε αυτά τα πράγματα Δεν ξέρω, καλύτερα, δηλαδή το αντιλαμβάνομαι περισσότερο να πείτε ότι έχετε μια συναισθηματική αντίδραση, αλλά παραδεχτείτε το. Δεν σας αρέσουν οι γενικά τροποποιημένοι οργανισμοί, ε, καλώ. α, μην Μα λέτε τώρα εδώ πέρα ψευδοεπιστημονικές ε, τέτοιε προτάσει Και συμφωνώ εδώ με τον κύριο Φιέλνερ. Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι έχουμε επιστημονικά στοιχεία, επιστημονική συνένεση όσον αφορά την χρήση των ε, προϊόντων όπως έχουμε και για την κλιματική αλλαγή. Και δεν είναι σωστό ε, για τους βουλευτές να δέχονται τα επιστημονικά στοιχεία μόνο για το ένα και όχι για το άλλο. Ε, είναι κάπως γελίο. Οπότε εγώ δεν θα υπερσφίσω αυτές τις αντιρρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο στην Κομισιόν στον κύριο Μπέρεντ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω πως έχω έρθει να αντικαταστήσω τον συνάδελφο που είναι επικεφαλής της ομάδας για τη βιοτεχνολογία και την ασφάλεια των τροφίμων, ο οποίος δυστυχώς ασθένησε και σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να ε, μιλήσουμε για αυτά τα σχέδια αντιρρήσεων. Όπως είπατε και εσείς, αυτές οι τρεις αιτήσει είναι για τη χρήση σε ε, τρόφιμα και ζωοτροφές ε, γενετικά τροποποιημένο ραβόστο και όχι για την καλλιέργεια. Στα διαδικαστικά να σας πω πως ακολουθήσαμε κατά γράμμα α, ε, ε, οδηγίες και κάναμε μια πολύ καλή αξιολόγηση κινδύνου στην ΕΦΣΑ. Τα αποτελέσματα είναι θετικά. Ε, για τους αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον. Για τις αντιρρήσεις που υπάρχουν για την αξιολόγηση κινδύνου της ΕΦΣΑ, να τονίσω πως εμείς κάναμε την αξιολόγηση κινδύνου, η ΕΦΣΑ μάλλον, σύμφωνα με τα όσα υπάρχουν στον 1829 του 2003 και τον εφαρμοστικό κανονισμό 503 του 2013 και σύμφωνα και με την σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Τα σχόλια των κρατών μελών για την εφαρμογή λήφθησαν πλήρω υπόψη από την ΕΦΣΑ κατά τη διάρκεια τη αξιολόγηση. Η ΕΦΣΑ ζήτησε να απαντηθούν όλε οι απαραίτητε ερωτήσει, έχει συλλέξει όλε τι απαραίτητε προφορίε από του ετούντε και για να αξιολογήσει αυτού του γενετικά τροποποιημένου ε, οργανισμού ε, ε, έκανε όλα τα απαραίτητα. Για την αντίρρηση και την έκθεση μειοψηφία από το ένα μέλος αυτό πρέπει να σας πω πως έτσι εξασφαλίζουμε την ακαιρεότητα της επιστημονική πραγματογνωμοσύνης, έτσι εργάζεται το πάνελ και αυτή η έκφραση της μειοψηφία δεν έχει να κάνει με ε, ε, το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά τις τρεις, τους τρεις υποσυνδυασμούς για τους οποίους έχει παραχθεί αυτή η η, έκθεση και αυτό έχει να κάνει ε, με τον αραβόστο σε στίβες. Η ΕΦΣΑ δεν δέχτηκε αυτή την ε, μειοψηφία, την άποψη μειοψηφίας και είπε πως αυτές οι τρεις υποκατηγορίες είναι ασφαλείς ε, βασιζόμενοι στην σόρευση σε που γίνεται με το συνδυασμό όλων των πρωτεϊνών σύμφωνα και μετά τα όσα έχουμε στην τεκμηρίευση. Λάβαμε και δημόσια σχόλια ε, κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας διαβούλευσης που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασιζόμενοι σε όλα αυτά προτείνουμε στα κράτη-μέλη να εγκρίνουν αυτούς τους τρεις αραβόστους προς εισαγωγή. Το σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης ευθυγραμμίζεται με τον 18-29 του 2013 και με τον κωδικό, και τον κώδικα για την ασφάλεια των τροφίμων, ε, για το περιβάλλον, για τα συμφέροντα του καταναλωτή και την ασφάλεια των ε, ζώων ε, όταν χρησιμοποιούνται γενικώ τροποποιημένοι οργανισμοί και λάβαμε τις εξή αποφάσεις που είναι αυτές που γνωρίζετε που ψηφίστηκαν στις 14 Ιανουαρίου στην Μόνιμη Επιτροπή χωρίς να εκδοθεί απόφαση λόγω πολιτικών κυρίως θεμάτων ε, και όχι λόγω επιστημονικών δεδομένων. Σύμφωνα με την Επιτροπολογία, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σχέδιο απόφαση στην Επιτροπή Ενστάσεων στι 22 Φεβρουαρίου. Σχετικά με τι ανησυχίε για, για τα προϊόντα αυτά τα φυτοπροστατευτικά, ε, στα οποία ε, υπάρχει ανοχή, και για τα μέγιστα όρια. Πρέπει να σας πω ότι λάβαμε υπόψη την την αντίστοιχη νομοθεσία, όπως αυτό καταγράφηκε και από κάποια μέλη εδώ του Κοινοβουλίου και πρέπει να σας πω πως οι γενετικώς τροποποιημένοι θα πρέπει αυτά τα μέγιστα ε, όρια καταλήπουν να τα ε, σέβονται ε, και να μην επιτρέπουν γλυφοσυνάτη, για παράδειγμα, που δεν επιτρέπεται. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την έγκριση του ζυζανιοκτώνου και δεν έχει να κάνει με τα μέγιστα όρια. Οπότε για τις παρατηρήσεις που έγιναν πως τα κατάλοιπα γλυφοσάτης και γλυφοσινάτης ε, στον αραβόστο δεν παρακολουθούνται, πρέπει να σας επιβεβαιώσω πως, δεν, πως αυτοί οι συνδυασμοί δεν αποτελούν τμήμα του προγράμματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ο αραβόστος δεν είναι στην κατηγορία των 13 πιο συχνά καταναλούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων, αλλά έχουμε πει στα κράτη-μέλη αν επιθυμούν στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου να τα συμπεριλάβουν, γιατί τα εθνικά προγράμματα προγράμματα συμπληρώνουν το κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου. Να σας πω τώρα ποια είναι η ενδεχόμενη επιρροή αυτών των ζυναζενιοκτώνων ε, και πώς λαμβάνεται υπόψη γιατί ε, ξέρετε πως οι καλλιέργειες αυτές ψεκάζονται με αυτά τα γενετικά τροποποιημένα ζανιοκτώνα και υπάρχουν κάποια ε, φαινοτυπικά και γεωπονικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Όταν λοιπόν προκύπτουν τέτοιου είδους αλλαγές και τροποποιήσεις ζητάμε να γίνουν κατά περίπτωση οι κατάλληλε μελέτες και αξιολόγηση κινδύνου. Για την καλλιέργεια σε τρίτες χώρες και τα κατάλληλα ζανιοκτώνων στα εμπορικά προϊόντα που προκύπτουν από αυτά η απόφαση να ελεγχθεί, με συγχωρείτε, να ε, ε επιτραπεί η καλλιέργεια είναι κυρίαρχο δικαίωμα αυτών των κρατών μελών και δεν μπορεί να επηρεαστεί από το κοινοτικό δίκαιο. Για την αναστολή του σχεδίου απόφαση μέχρι η διαδικασία αντίρρηση έχει ε, περατωθεί, εμείς καταθέσαμε πρόταση που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να περιορίσουν τις αγωγέ αυτών των τροφίμων και ζωοτροφών στη χώρα τους. Αυτή η πρόταση απερίφθη από το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό, και περιμένουμε να συνεχίσουν οι συζητήσεις με το Συμβούλιο για να δούμε τι θα αποσυστεί. Εμείς ε, έχουμε μια καταθέσει μια φιλόδοξη πρόταση για ε, να έχουμε περισσότερη διαφάνεια στην αξιολόγηση κινδύνου της ΕΦΣΑ και με το Κοινοβούλιο καταλήξαμε σε μια πρώτη συμφωνία όπου ελπίζουμε θα εγκριθεί τις επόμενες εβδομάδες. Εν κατακλείδη λοιπόν να πω πως Υπογραμμίζω πω δεν υπάρχει κανένα λόγο στο σχέδιο αυτό απόφαση να αποσυρθεί, μια και όλε οι διαδικασίε που υπάρχουν στο σχετικό κανονισμό έγιναν ε, σεβαστέ και οι εφαρμοστικέ εξουσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σεβαστέ καθ' όλη τη διαδικασία. Τέλο, το δικαίωμα εξέταση του Κοινοβουλίου περιορίζεται στο θέμα του κατά πόσο το σχέδιο αυτό ξεπερνά τι εφαρμοστικέ ε, εξουσίε που έχουμε στο ε, βασικό κείμενο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη αυτό το να το ε, υποβάλει προσέγγιση πέραν του σημείου στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Ενημερώνω την Επιτροπή ότι θα ψηφίσουμε αυτές τις αντιρρήσεις αργότερα σήμερα, σε μια μισή ώρα περίπου. Και αναμένουμε να εγκριθούν ε, στην Επιτροπή και στην πρώτη Ολομέλεια του Μαρτίου. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι μια άλλη αντίρρηση για τις δραστικές ουσίες ε, συμπεριλαμβανομένης της διαλκοπρίν. Για το Θεακλοπρίν, δίνω το λόγο ε, στην εισηγήτρια την κυρία Σιλβί Κοντίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Θεακλοπρίν είναι νοικοτινοειδές που χρησιμοποιείται στην εντατική γεωργία ευθύνεται για την αύξηση της νησιμότητας των επικονιαστών και των μελισσών. Η ουσία αυτή είναι ολοένα και πιο ανησυχητική. Η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν απαγορεύσει την χρήση. Ωστόσο, η Κομισιόν αποφάσισε χωρίς τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρατείνει κατά ένα έτος την άδεια κυκλοφορίας του με τις επιδράσεις που έχει αυτό στις μέλισσες. Είχε δοθεί άδεια για 10 χρόνια και εδώ και 4 ε, χρόνια η ΕΦΣΑ την ε, επανεξετάζει. Αυτή η επανεξέταση θα παραταθεί κατά ένα έτος πριν δημοσιευτούν τα συμπεράσματα για αυτή την ουσία της οποίας ε, η επιβλαβής δράση έχει ήδη εντοπιστεί από τη Γαλλία και το Βέλγιο, δύο κράτη-μέλη. Ακόμα χειρότερα αυτή η απόφαση λαμβάνεται πριν καν δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη γνωμοδότησή του για αυτή την άδεια κυκλοφορία, διότι η δική μα γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική. Πράγματι, η Κομισιόν έχει ήδη δημοσιεύσει αυτή την παράταση τη ε, αδειοδότηση σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Δίνει την άδεια δηλαδή κυκλοφορία μια δραστική ουσία κατά τη γνωμοδότηση ενό δημοκρατικά εκλεγμένου κοινοβουλίου, σε περίπτωση που υιοθετηθεί η δική μα ε, ένσταση στη σκανδαλώδη. Αυτή η κατάσταση προστίθεται ε, αυτή η συμπεριφορά της Κομισιόν όσον αφορά τη βιοπικιλότητα και ένα έτος ακόμα ε, άδικο για τους Γάλλους και Βέλγους αγρότες οι οποίοι αντίθετα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρησιμοποιούν πλέον αυτές τις ουσίες. Έτσι λοιπόν η ε, γεωργοί στη Γαλλία και το Βέλγιο όπου η ουσία έχει απαγορευτεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 δεν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν αλλά θα συνεχίσουν να υφίστανται τις ε, εισαγωγές από το εξωτερικό γεωργικών προϊόντων που έχουν περιέχουν αυτό το νοικοτενοειδέ που είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες. Γι' αυτό το λόγο ζητώ από τους συναδέλφους μου να υποστηρίξουν αυτή την αντίρρηση που ε, υπέβαλαν πέντε πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο μιλητής από τους σοσιαλιστές, η κυρία Κάντεμπαχ, έχετε το λόγο. Α τα πούμε απλά λοιπόν αυτή τη φορά. Συμφωνώ πλήρω με την πρόλαβή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ρίς, λοιπόν, από την Άλντε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η αντίρρηση που υποβάλλουμε ε, αντιτίθεται στην επέκταση της άδεια ε, του θεαλκοπρίντα, που είναι αυτό το οικοτινοειδές και που σκοτώνει τις μέλισσες όπως γνωρίζουμε. Τρίτη παράταση σε τρία χρόνια χωρίς καμία ανάλυση στην πραγματικότητα όσον αφορά τι βλάβε που προκαλεί διότι μόνο η ανανέωση απαιτεί τέτοιε αναλύσει, Ωστόσο, οι επιστημονικές έρευνες ε, έχουν εξελιχθεί, ε, έχουν αλλάξει τα πορίσματα μετά το 2005 όταν ε, δόθηκε άδεια τέτοια, για αυτή την ουσία στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Ε, κυταροτοξική, γονιδιοτοξική, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Ζυζανιοκτώνων ε, τη χαρακτηρίζει ως ε, ενδοκρινικό διαταράκτη, λένε ότι είναι καρκινογόνος, τοξική για την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Παρόλα αυτά, η... και ο Γαλλικό Οργανισμός για την Υγεία και το Περιβάλλον σε μία έκθεση του Μαΐου του 2018 ζήτησε μείωση της χρήση στο μέγιστο λόγω του επικίνδυνου χαρακτήρα τη ουσία και έγινε, όπω είπαμε, στη Γαλλία, στη Γαλλία και εδώ ε, πέρσι το Σεπτέμβριο μετά από τον ε, Ιούνιο όπου η Βαλονία και οι Βρυξέλλες ε, επέβαλαν την απαγόρευση. Τα κείμενα είναι σαφές. Το θέμα είναι να προστατεύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και το περιβάλλον μας. Αυτή η αντίρρηση θα έλεγα είναι ακριβώς αυτό. Δεν, δεν, δεν υπάρχει καμία δεν δημιουργεί καμία αμφιβολία. Δεν καταλαβαίνουμε πώ συνεχίζεται να επιτρέπεται η χρήση μια τόσο καταστρεπτική ουσία. Δεν θέλουμε να στέλνουμε τέτοιο μήνυμα στου Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο τώρα ξανά. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Στην Επιτροπή. Κύριε Μερέντ. Yes. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ο κανονισμός, στον οποίο αναφέρεται εδώ το σχέδιο αντίρρησης, έχει ήδη εγκριθεί στις 31 Ιανουαρίου, δημοσιεύτηκε στις 5 Φεβρουαρίου, 2019 καθώς 169 επεκτείνει την περίοδο έγκρισης 42 ουσιών για τις οποίες εξέπνευσε η έγκριση μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 30 Απριλίου 2019 ε, κατά ένα έτος. Οι παρατάσεις αυτές είναι αναγκαίες γιατί, με συγχωρείτε κύριε Μπέρεντ, Υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Η κυρία Γκέρλινγκ ε, θέλει να ζητήσει τον λόγο. Οπότε θα δώσω τον λόγο στην κυρία Γκέρλινγκ πρώτα. Και μετά μπορούμε να επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει κύριε Γκέρλινγκ. Ε, ευχαριστώ, ναι. Ε, παίρνω τον λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ που δεν υποστήριξε αυτήν την αντίρρηση και δεν θα την υποστηρίξει, θα είμαι σύντομη, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί αυτό. Γιατί δεν υπάρχει ομοφωνία εδώ. Θα ήθελα απλώς να πω ότι η λέξη νεονικοτινοειδή σαφώς έχει κάποια κάποιες αρνητικές εικόνες ε, που φέρνει στο μυαλό, αλλά θα πρέπει να δείτε τις ουσίες ε, που καλούνται νεονοικοτινοειδείς, γιατί είναι διαφορετικές, χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο και λειτουργούν διαφορετικά, οπότε η συγκεκριμένη ε, δεν χρειάζεται βασικά σε αυτή την αντίρρηση να συζητήσουμε το ε, ναι ή όχι. Νομίζω η κυρία Γκοντάν θα πρέπει να αντιληφθεί το σύστημα πριν αρχίσει να μιλάει τόσο πολύ στην Επιτροπή. Πρόκειται για αντίρρηση σε εφαρμοστική πράξη, οπότε το θέμα δεν είναι ε, το εάν αγνοείται το Κοινοβούλιο, αλλά να αντιληφθούμε πώ λειτουργεί το Κοινοβούλιο και ποιο είναι ο ρόλος μας στην διαδικασία. Και στην περίπτωση αυτή, ξεκάθαρα, το θέμα είναι ότι η ανανέωση δεν έλαβε χώρα λόγω του συστήματος που έχουμε αναγνωρίσει. Έχουμε και τον νόμο περί ζανιοκτώνων και τη Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα που αναγνωρίζουν ότι δεν λειτουργεί καλά το σύστημα. Τώρα θα εγκρίνουμε ένα νέο σύστημα με το νέο Γενικό Νόμο για τα Τρόφιμα. Οπότε ελπίζουμε να ξεπεραστεί αυτό το μπλοκάρισμα. Οπότε ουσιαστικά λέμε μόνο το προϊόν αυτό έχει καθυστερήσει χωρίς να φταίνει οι κατασκευαστές και σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού που λέει όταν για λόγους πέραν του ελέγχου του ετούντος θα εκπνεύσει η προθεσμία τότε έχουν δικαίωμα σε παράταση. Αυτό είναι όλο. Δεν ζητάνε άλλα 10 χρόνια. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι θα θέλαμε να γίνει αυτή η αναθεώρηση αλλά πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που θα μας επιτρέπει να λαμβάνουμε αυτή την απόφαση. Και το γεγονός ότι το Βέλγιο και η Γαλλία το απαγόρευσαν και πάλι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το απαγορεύσουμε όλοι. Μπορεί να έχουν τους δικούς τους λόγους, εσωτερικούς πολιτικούς. Ε, λογικό είναι να έχουμε κάποια αντίρρηση, να τεθεί ενισχύ το νέο σύστημα και να υπάρξει σωστή ανανέωση αυτού του προϊόντος. Σας ευχαριστώ. Επανερχόμαστε στην Κομισιόν λοιπόν. Συνεχίστε από εκεί που σας διακόψαμε και μας συγχωρείτε. Νομίζω ακούσαμε αυτά τα οποία είπατε. Μπορείτε να συνεχίσετε την παρουσίασή σας. Έχετε τον λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ε, μπορώ να είμαι πιο σύντομο τώρα, γιατί η κυρία Γκέρλινγκ ε, είπε πολλά από αυτά τα οποία είχα να πω. Και το βασικό είναι ότι πρόκειται πράγματι για μια, ε, μια παράταση για καθαρά διοικητικούς λόγους. Δεν πρόκειται για επανεξέταση του φακέλου που σχετίζεται με την ανανέωση της έγκρισης της ουσίας και όπως σωστά σημείωσε η κυρία Γκέρλινγκ, το άρθρο 17 του κανονισμού 1107 του 2009 υποχρεώνει την Κομισιόν να επεκτείνει την περίοδο έγκρισης για ουσίες για τις οποίες δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης ε, για λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχο του ετούντος. Και αυτό συμβαίνει εδώ. Να υπογραμμίσω ότι στο σύστημα που έχουμε πρώτα απ' όλα το κράτος μέλος κάνει μια αξιολόγηση της αίτησης ανανέωσης, την υποβάλλει στην ΕΦΣΑ για μια διαδικασία ελέγχου και μετά μπορεί η Κομισιόν να λάβει απόφαση. Στην περίπτωση αυτή το κράτος μέλος καθυστέρησε 24 μήνες στο να δώσει την έκθεση αξιολόγησης και η ΕΦΣΑ μετά άλλους 4 μήνες πριν βγάλει τα συμπεράσματα της. Ε, αυτά λοιπόν δεν οφείλονται στον Ετούντα, οπότε οι λόγοι για την καθυστέρηση είναι πέρα τον ελεγχό του. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 17, η Καμψιόν δεν είχε άλλη, άλλη επιλογή παρά να παρατείνει την ε, έγκριση της ουσίας. Η κυρία Ρίς αναφέρθηκε στην κατάταξη, αλλά και πάλι το άρθρο 17 δεν κάνει διάκριση μεταξύ ουσιών που πληρούν κάποιες κατατάξεις ή όχι. Η υποχρέωση παράτασης παραταση ειναι γενική και ισχύει για όλες τις ουσίες. Επιπλέον το σχέδιο ψηφίσματος λέει ότι ο κανονισμός που επεκτείνει την έγκριση υπερβαίνει τις εφαρμοστικές αρμοδιότητες κομισιών. Όχι. Αντιθέτως, όπως εξήγησε το άρθρο 17 του κανονισμού μας υποχρεώνει να το κάνουμε και αν δεν το είχαμε κάνει θα είχαμε υπερβεί τις εφαρμοστικές αρμοδιότητές μας. Τέλος, να σας ενημερώσω ότι ο φάκελος, τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ και η αξιολόγηση του κράτους μέλους έχουν φτάσει στην Κομισιόν στις 22 Ιανουαρίου και άρα ξεκινάει η διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ανανέωση και αναμένουμε να παρουσιαστεί μια απόφαση τον επόμενο μήνα αλλά όχι πριν της 30 Απριλίου. Γι' αυτό απαιτήθηκε αυτή η παράταση. Ελπίζουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί και αν η απόφαση είναι για μία ανανέωση τότε βεβαίως η παράταση θα ανακληθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν θα ψηφίσουμε σήμερα για τις αντιρρήσεις αυτές και αν ε, περάσουν από εμάς θα πάμε στην ε, Ολομέλεια στην πρώτη του Μαρτίου και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Εδώ έχουμε ακόμα μία αντίρρηση. Είναι μία αντίρρηση σύμφωνα ε, με ε, τα του κανονισμού για ουσίες όπως η κλωθιανιδίνη. Θα δώσω λοιπόν πρώτα στους εισηγητές και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μαντάμ Ντελαέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όντως και πάλι έχουμε ε, κοτινοειδές, αλλά αυτή τη στιγμή έχει να κάνει ε, με το μέγιστο όριο. Και αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση, μια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ουσία αυτή ε, απαγορεύεται χωρίς καμία καμία εξαίρεση παρά μόνο σε θερμοκήπια αν οι σπόροι δεν ξεφύγουν από την περίφραξη του θερμοκηπίου. Αλλά απαγορεύεται στα ε, χωράφια ε, έξω. Οπότε γιατί περνάμε από το 0,03 στο 0,3 μιλιγκράμμ το κιλό. Μου φαίνεται πως αυτό είναι μια αύξηση ε, μία μελιτέα και περιμένω ε, να μου δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγήσεις για το πώς και γιατί οι Ευρωπαίοι Γεωργοί που ε, εμπίπτουν σε αυτό τον κανόνα θα πρέπει να αλλάξουν παρόλο που το έχουν παραδεχτεί, παρόλο που λειτουργεί και πώς θα αιτιολογήσουν αυτή την αύξηση. Εγώ είμαι κατά. Πολύ στεναρά κατά παρόλο που η διαδικασία έχει γίνει σεβαστή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μένα δεν είναι διαδικαστικό το θέμα, είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα ουσιαστικό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν να είναι πιο προστατευμένοι και δεν νομίζω ότι αυξάνοντας έτσι αυτό το όριο σε ένα νέο νοικοτινοειδές θα εξασφαλίσουμε πως ο Ευρωπαίος πολίτης θα αισθάνεται πιο ασφαλής και θα αισθάνεται πως με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε την υγεία του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάντεμπαχ. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Ακούστηκαν ήδη, εφόσον είναι κοινή αντίρρηση Μα δεν έχω να προσθέσω κάτι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρίς, λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι αυτή ήταν η δεύτερη αντίρρηση στην οποία συμπροεδρεύω, για να το πω έτσι, σήμερα το πρωί. Η επιχειρηματολογία είναι ουσιαστικά ίδια. Θέλω να απαντήσω στην κυρία Γκίρλινγκ και στα επιχειρήματα τη Επιτροπής όσον αφορά τα διαδικαστικά. Εγώ γνωρίζω τη διαδικασία, αλλά το θέμα δεν είναι διαδικαστικό εδώ μόνο. Γνωρίζουμε και την κατάσταση του πληθυσμού των μελισσών ε, στην Ευρώπη, παγκοσμίω, ε, τι ε, διάφορε απόψει μα για το θέμα και παρατηρούμε και πώ εξελίσσονται τα πορίσματα τη επιστήμη. Εμεί θέλουμε λοιπόν να υπόλοιπα αντίρρηση παρότι δεν έχουμε αρμοδιότητα γνωμοδότηση, για να το πω έτσι αυτό των νοικοτινοειδές ε, η κλωθιανιδίνη η Κομισιόν μας προτείνει να δεκαπλασιάσουμε το μέγιστο όριο καταλήπων που θα επιτρέπεται ενώ η ουσία είναι υψηλατοξική ειδικότερα για τις μέλισσες με βλαβερές συνέπειες γνωστές μάλιστα λόγω της χρήσης ε, η οποία έχει απαγορευτεί ε, στα χωράφια και περιορίζεται στην Ευρώπη από το 2013. Ο Καναδάς συνεχίζει να τη χρησιμοποιεί την ουσία και ζητάμε να ανεβάσουμε, να δεκαπλασιάσουμε το όριο, ώστε να μπορεί ο Καναδά να μα στείλει τι πατάτε του. Αυτό γίνεται. Δεν ζητάω, από την Κομισιόν να το επιβεβαιώσω, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα. Δεν πρόκειται εμεί να πάμε να υπαγορεύσουμε νομοθεσία στο εταίρο μα στον Καναδά, αλλά ούτε μπορούμε να κάμπτουμε εμεί τι δικέ μα νομοθεσίε και τα πρότυπά μα. η περιεκτικότητα αυτή παγιώθηκε όταν έγινε η συμφωνία για το ΣΕΤΑ ε, και με τρόπο μετακίνητο. Ε, είναι λίγο φυσικά περιττό το ότι έχουμε αυτό το όριο γιατί απαγορεύεται αυτή η ουσία σε εμά. Παρ' όλα αυτά δεν πάμε να αποτελεί υποβάθμιση των προτύπων μα και των αξιών μα ε, κάτι τέτοιο. Μα λένε ότι είναι τόσο βλαβερή η ουσία που την απαγορεύουμε. Τι νόημα έχει λοιπόν να χαμηλώσουμε τα πρότυπά μα και τα οριά μα ώστε να ενθαρρύνουμε de facto τη συνέχιση τη χρήση αλλού ουσιαστικά, όχι απλά ε, κάνουμε σαν να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ε, κάτι άλλο τώρα, υπάρχει λόγος ε, να, για να το ε, για να αναφερθώ και σε κάτι διαφορετικό, υπάρχει λόγο να μα στέλνουν πατάτε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ουσιαστικά, όπω είπε και η κυρία Κάτεμπαχ, εν συντομία δεν το θέλουμε. Φέρουμε αντίρρηση. Και τέλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενη εισηγήτρια, κυρία Κοντίν. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπουμε ακριβώς τι απέσια αποτελέσματα έχουν αυτές οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Έχουμε τους κανόνες του Καναδά, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την οικονομία, ούτε για μας να τους επιβάλλουμε εδώ. Η κλωστιαδίνη απαγορεύεται. Πολύ σωστά άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι νεονικοτονοειδές που επηρεάζει πολύ αρνητικά τους επικονιαστές. Και εσείς λέτε να πολλαπλάσουμε επί 10 τα μέγιστα όρια στις πατάτες που εισάγουμε τον Καναδά. Τρία σημεία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πρώτα, αυτή η αύξηση των ορίων δεν ανταποκρίνεται στα όσα θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως δέσμευση για τους επικονιαστές. την ίδια συνέπεια είχε την καταστροφή των ε, μελισσών στη Βόρεια Αμερική που είχαμε δει και εδώ έχουμε περιβαλλοντολογικές ευθύνες. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε ως υπεργολαβία αυτές τις κακές πρακτικές που ήταν καταστροφικές για το περιβάλλον στους φίλους Καναδούς. Δεύτερον, ανθρώπινη ανθρώπινη υγεία. Αυτή η αύξηση των καταλήπων στα τρόφιμα είναι απαράδεκτη. Και βλέπετε όλοι πως υπάρχουν μελέτες επιστημονικές, λεπτομερείς που έδειξαν πόσο τοξικό είναι αυτό το προϊόν, αυτή η ουσία. Ακόμα χειρότερο, η αξιολόγηση της ΕΦΣΑ μιλά για τις συνέπειες που έχει ε, Ιδίω όταν συνδυάζεται με άλλες βλαβερές ουσίες όπως την ηθικοτέλεια ε, που είναι χημική βόμβα όταν βρίσκεται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Τέλος, η έκθεση αυτή η πρόταση αυτή της Κομισιόν ανοίγει το δρόμο για τον αθέμητο ανταγωνισμό με τους Ευρωπαίους γεωργούς που δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν αυτή την ουσία, που με τον τρόπο αυτό δεν έχουν τρόπο ε, ελέγχου των ζιζανιών ε, και των εντόμων, ε, ενώ θα τον έχουν οι Καναδοί από τους οποίους θα εισάγουμε. Και είναι φρικτό για το περιβάλλον και δεν θα δώσει καλά αποτελέσματα, γιατί οι ευρωπαϊκές πατάτες τελικά θα υποκύψουν στον ε, ανταγωνισμό των δηλητηριασμένων και φθηνών πατατών από τον Καναδά. Ευχαριστώ μετά από αυτό το γύρο ομιλητών. Δίνω το λόγο στα άλλα μέλη τη ε, Επιτροπή, την κυρία Γκέρλεγκ. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπε τρει. Θέλω να σας αποδείξω λοιπόν ε, πώς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία. Θα ρωτήσω λοιπόν κάτι στην Κομισιόν το μέγιστο όριο καταλήπων, το MRL, όταν ορίζεται για μια ουσία και ειδικότερα για ουσίες απαγορευμένες για, τη, για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που μπορεί να είναι παρούσε σε πολύ μικρές ε, περιεκτικότητες ε, εισαγόμενα προϊόντα και το τονίζω, πολύ μικρές περιεκτικότητες εξορισμού το MRL είναι κατάλοιπο και συνεπώ μικρή ποσότητα, το, η λέξη κατάλοιπο υπενήστε μικρή ποσότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι υπερβολικά δυσανάλογες οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι ε, συναδελφοί για δηλητηριώδη προϊόντα που εισάγουμε. Τα MRL ακριβώς αυτό προλαμβάνουν. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο αναλογικοί και στη γλώσσα μα εδώ. Είναι υπερβολές αυτά που ακούμε. Αλλά Θέλω να ρωτήσω το εξή. Για να υπάρχει μέγιστο όριο καταλήπων για μια τέτοια ουσία, αυτό ορίζεται από την ΕΦΣΑ μέσω μια διαδικασία η οποία είναι αυστηρή και βασίζεται στις τοξικολογικές επιδράσεις στον τελικό χρήστη του προϊόντος ή το επίπεδο αυτό ορίζεται δυνάμει του κάποιου προτύπου εμπορικού που έχουμε. Ουσιαστικά πόσο τεκμηριώνεται επιστημονικά, γιατί ε, εδώ υπάρχει πιθανότητα να το δεκαπλασιάζουμε και να μην έχουμε ε, απίδραση στον άνθρωπο. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα. Και αυτό που ρωτάω την Κομισιόν λοιπόν ξανά είναι πώ ορίζεται αυτό το MRL και πώ καταλήγεται στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεκαπλασιάσετε το όριο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Φλόρεντς. Ευχαριστώ που μου δίνετε πάλι την ευκαιρία. Κοιτάξτε, τα νεονικοτινοειδή, ε, τι να σας πω, είναι λίγο κοινοβιστικά, δεν θα μας σκοτώσουν αύριο. Ε, ακούω για απαγορεύσεις. Ε, κοιτάω εδώ πέρα τους ε, κυρίους Κομισιόν. Ε, δεν μπορείτε να επιβάλλετε τους κανόνες, τους ευρωπαϊκούς. Είστε οι θεματοφύλακες συνθήκης. Δευτέρα στη ε, εργοστάσιο της Ζάχαρης ε, το δικό μου ήρθαν 2.000 αγρότες και μου λένε ότι η Ευρώπη θα απαγορεύσει τα νεονικοτινοειδή και στη γειτονιά μας 18 χώρες θα κάνουν εξαίρεση και η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα. Ο κύριος Γιούνκερ έγραψε μάλιστα σε ένα άρθρο και λέει ότι ε, έχω βαρεθεί να παίζω ε, το παιχνίδι αυτό στην Ευρώπη. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Έχουμε ένα νόμο ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί. Οι αγρότες έχουν μείνει ταπεί. Λοιπόν, και τα χωράφια επίσης είναι νεκρά. Όποιος βρει μικροοργανισμούς να του κάνω το τραπέζι. Κοιτάξτε, μιλάμε για τρεις καρπούς ε, εδώ πέρα και η Κομισιόν μιλάει για το εάν θα κάνει έγκριση για την ε, οικιακή χρήση. Μιλάμε για καταστροφή. Όχι, ε, απαγόρευση σημαίνει απαγόρευση. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε συνεχώς να, βάζουμε ερωτηματικά, ας τα παρατήσουμε και στις εκλογές. Όχι, σταματήστε τη χρήση είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στη Γεωργία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τον λόγο έχει πάλι η Κομισιόν ο κύριος Μπέρεντ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε να πω ότι το σχέδιο αυτό αφορά το να ορίσουμε MRL και δεν σχετίζεται με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλόρενς ε, στην παρέμβασή του, δηλαδή την έγκριση κάποιων προϊόντων, η δραστική ουσία των οποίων απαγορεύεται από κατεπίγουσες παρεκκλήσεις που έδωσαν τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι απολύτω αρμοδιότητα των κρατών και κομισιών, όπως και εσείς. Λυπάτε για το ότι το χρησιμοποιούν τόσο πολύ τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό δεν ε, σχετίζεται με το σχέδιο κανονισμού εδώ πέρα. Λοιπόν, πολλοί ομιλητέ ε, αναφέρθηκαν στους κινδύνους ε, που περιέχουν αυτά για τις ε, μέλισσες και το περιβάλλον. Και πράγματι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίσει την χρήση τους μόνο σε θερμοκήπια και όχι στην Ήπεθρο. Οπότε το θέμα των μελισσών το έχουμε αντιμετωπίσει πλήρως ε, στην αδειοδότηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό το οποίο προτείνουμε εδώ πέρα αφορά εισαγωγές από άλλες χώρες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Καναδάς, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, μπορεί να παρέμβει στην νομοθεσία και την αδειοδότηση τρίτων χωρών. Είναι κυρίαρχη απόφαση αυτών των χωρών και δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε ε, να δώσουν άδεια σε προϊόντα ε, επειδή απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός αυτός ε, ασχολείται μόνο με τον αντίκτυπο στην υγεία των καταναλωτών. Αυτό για να απαντήσω συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας Γκέρλινγκ έχει αξιολογηθεί σε μια διαδικασία δύο φάσεων, πρώτα από ένα κράτος και μετά από την ΕΨΑ με βάση διεθνείς μεθοδολογίες και αξιολόγηση κινδύνου που εφαρμόζει ΕΦΣΑ. Όσον αφορά το πακέτο των δεδομένων περί τοξικολογίας. Οπότε η ΕΦΣΑ έχει επιβεβαιώσει ότι το MRL για τις ουσίες αυτές τις ε, πατάτες ε, τα κατάλοιπα δηλαδή είναι ασφαλή για τους καταναλωτές. Να υπογραμμίσω επίσης πως η Κομισιόν δρά εντός ε, των αρμοδιοτήτων που έχει σύμφωνα με τον οργανισμό 396-2005, το άρθρο 14 συγκεκριμένα που υποχρεώνει την Κομισιόν να υποβάλει ένα σχέδιο κανονισμού εντό τριών μηνών από την επιστημονική γνωμοδότηση τη ΕΦΣΑ, γνωμοδότηση η οποία βασίζεται στα άρθρα 6 έως 11 του κανονισμού. Οπότε το σχέδιο κανονισμού συμφωνεί με τις αρχές και τους στόχους του κανονισμού που είναι το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Και άρα και πάλι δεν βλέπουμε κάποιον λόγο να ανακαλέσουμε την πρόταση αυτή, καθώς συμμορφώνεται με τις προτάσεις και τους στόχους του κανονισμού και στόχο έχει μόνο την προστασία της ανθρώπινης υγείας, συγκεκριμένα των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τον λόγο έχει η κυρία Ντελαή και ο κύριος Φλόρεντς. Δεν θα ξανανοίξω τώρα την συζήτηση αν έχετε κάποια πολύ σύντομη ερώτηση προς την Κομισιόν, να σας δώσω τον λόγο για να υπάρξει κάποια διευκρίνηση. Και μετά θα ξαναδώσω τον λόγο στην Κομισιόν για να αντιδράσει και μετά τέλος. Η κυρία Ντελαή. Δεν θα ξανανοίξω τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Θέλω απλώς να καταγραφεί η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δείχνει και αποδεικνύει πως αυτό το αίτημα για αύξηση απλώς ανταποκρίνεται σε ένα πρόβλημα εμπορικής συμφωνίας. Εγώ είμαι κατά. Και δεν είναι μία απόκριση που δέχονται σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες από μια Ευρώπη που πρέπει να τους προστατεύσει και δεν είναι με αυτά τα επιχειρήματα που θα συμφιλιώσουμε τους Ευρωπαίους με το ευρωπαϊκό project. Κύριε Φλόρενς. Τώρα, κοίταξε, ε, δεν θέλω να κατηγορώ εδώ πέρα τον άνθρωπο της Κομισιόν. Όταν συζητήσαμε όμως τα θέματα των νέων οικοτινοειδών, κινηθήκαμε σχετικά γρήγορα. Και μετά ήρθαν οι αγαπητοί μας φίλοι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν κάναν το ίδιο. Και τι έκανε η Κομισιόν, είπε ναι το Συμβούλιο δεν θέλει, το Κοινοβούλιο υπερβάλλει και γράφει μετά μια λεξούλα που λέγεται επικουρικότητα. Ο καθένας μπορεί να δώσει άδεια και ο άλλος ε, όχι. Αυτό είναι το λάθος σας. Πρέπει να σταματήσει αυτή η νοοτροπία όταν μιλάμε για υγεία. Ε, καλύτερα μην γράφουμε νόμους καθόλου. Αλλά ε, τι να σου πω, δηλαδή έχουμε 18 χώρες που θα χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα στις ε, πατάτες ε, και στα ζαχαρότευτλα, ειλικρινά σας λέω, εξοργίζει τους ε, αγρότες μου. Εσείς δεν ψηφίζεστε, εμείς πρέπει να ψηφιστούμε και θα μας γυρίσουν την πλάτη σας, το λέω. no, ναι, I really... Ναι, ναι, ε, εδώ όμως πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση, δίνω και πάλι τον λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο Μπέ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δεύτερη δυνατότητα που μου δώσετε να πάρω το λόγο. Σε σχέση με τα όσα είπατε, δεν έχει καμία σχέση αυτό που κάνουμε με την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Όχι, είναι οι κανόνες του σχετικού κανονισμού για τα ανώτατα όρια που λέει πως τα αιτήματα για την εισαγωγική ανοχή μπορούν να υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς και υπάρχει μια διαδικασία, ένα πακέτο δεδομένων και μια αξιολόγηση που προβλέπονται από τα κράτη-μέλη και από, τον, ε, από την ΕΦΣΑ. Δεν είναι κάτι που σχετίζεται με τις ελεύθερε συναλλαγέ είναι στον κανονισμό. Κύριε Φλόρεντς, συνεχίζω. Συμφωνήσαμε κι εμεί. πως δεν είναι αποδεκτή αυτή η διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων και εξαιρέσεων από τα κράτη-μέλη και έχουμε ζητήσει να τα αξιολογήσει η ΕΦΣΑ, να δούμε αν δικαιολογούνται σύμφωνα με το όσο έχουμε στον κανονισμό και η ΕΦΣΑ είπε πως για τα όσα εξέτασε τα 2 το, τα δύο τρίτα είναι αποδεκτά, το ένα τρίτο όχι και γι' αυτό για πρώτη φορά στο άμεσο μέλλον θα προτείνουμε για να μην ε, δίνουν τέτοιες επίγουσες εγκρίσεις στα ευρωπαϊκά, ε, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ε, ένα σχέδιο έτσι ώστε αυτό να αποφεύγεται. Καταλαβαίνω βέβαια το ότι το πρόβλημά σας έχει να κάνει με τα τέφτλα και όχι με τις πατάτες και την καλλιέργεια αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Θα το ψηφίσουμε σήμερα αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα αν ε, εγκριθεί η αντίρρηση θα πάει στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου για προσψήφιση. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 11.30, οπότε διακόπτουμε και θα σας παρακαλούσα να επιστρέψετε ακριβώς ε, στις 11.30 για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία στην ώρα της. Ευχαριστώ.

Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Καθίστε λοιπόν. Ελέγξτε τις κάρτες ψηφοφορίας σας, αν τις έχετε μαζί σας, αν τις έχετε βάλει στα μηχανήματα. Ελέγχουμε λοιπόν τις κάρτες πρώτα απ' όλα. Ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, πατήστε το οποιοδήποτε κουμπί. Μόλις ελέγχουμε. Για να δούμε αν έχουμε το σωστό αριθμό βουλευτών, να λειτουργούν σωστά όλα τα μηχανήματα, πέρα της ψηφοφορίας. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Πρώτο σημείο η προσωρινή ε, Συμφωνία για τη Διαφάνεια και τη Βιωσιμότητα τη Εξολόγηση Κινδύνου στην Αλυσίδα Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη Επόμενο σημείο, εδώ έχουμε πολλές ψήφους και αντιρρήσεις. Ε, ε, η πρώτη αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού Γενετικό τροποποιημένο αραβόστο 4114. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη πάλι αντίρρηση για τον γενετικό τροποποιημένο αραβόστο μον 87411. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη αντίρρηση. Η γενετικός τροποποιημένο αραβόσιτος BT11 και ούτω καθεξής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη αντίρρηση. Δραστικές ουσίες που περιέχουν θιακλοπρίντ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελευταία αντίρρηση για τα ανώτατα όρια καταλήπων ε, για την κλωθιανιδίνη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης συγκρίνεται. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Η στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού. Σχέδιο ψηφίσματος, σχέδιο πρώτας ψηφίσματος, συμβαστική 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ας τσεκάρουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 14. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο, η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 16. Συγγνώμη, είχατε δίκιο. Είχαμε διαφορετικέ ψήφου στο ΕΛΚΑ. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη για το λάθο. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 ε, θα ψηφιστεί επιπλέον υπέρ, κατά, αποχ... αποχές, εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Closes, uh, vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 98. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 98. Πέρας. Εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβεβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε τη 15, τροπολογία 15. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 100 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα 142 υπέρ κατά αποχές απορριπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά να ελέγξουμε την συμβιβαστική 16 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο. Η ίδια πλειοψηφία νομίζω να ελέγξουμε τη συμβιβαστική 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 188 188 πέρας απορρίπτεται συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 223 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 239 υπέρ καταπίπτει, συγγνώμη, συμβιβαστική 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 185 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 251 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 252, να ελέγξουμε τη 251 λοιπόν, ελέγχουμε τη 251, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.80 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά να το τσεκάρουμε 2.80 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 2.81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 269 δεύτερο τμήμα πρέπει να ψηφιστεί υπέρ κατά αποχές ας το τσεκάρουμε 269 δεύτερο τμήμα επιπροσθέτω στη συμβιβαστική 32 ε, πέρας ψηφοφορίας ε, απορρίπτεται 288 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 290 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 291 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.92 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.94 ε, καταπίπτει όχι πρέπει να ψηφιστεί 2.94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 308 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 309 υπέρ, κατά, αποχές. Να το τσεκάρουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, 309 πέρα εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 318 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 319 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε την 319. Να ελέγξουμε 319. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 320 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 322 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 324 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 325 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 337 υπέρ κα, κατά αποχές εγκρίνεται 3.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.56 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται να ελέγξουμε την 356. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καλά τα χέρια σας, γιατί μερικές φορές δεν φαίνεται καλά. Τι ψηφίζετε. 3,57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε όμως. 3.57 θα την ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβεστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 366 υπέρ. Κατά. Είναι υπέρ ή κατά τώρα αυτό. Α, είναι δική τροπολογία, συγγνώμη, ναι. Εγκρίνεται λοιπόν. 368 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει μετά. Συμβεστική 40 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 374 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 384 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 378 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 379 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 380 υπέρ Καταπίπτει, συγγνώμη. Ε, καταπίπτει και 381, 383. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεστική 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 392. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 394. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική 43. Υπέρ. Κατά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 κατά αποχές απορρίπτεται τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συγχαρητήρια για τον συνεισηγητή Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο Είναι η εποχιακή αλλαγή της ώρας και είναι ο φάκελος αυτός. Τροπολογία 4 που είναι απόρριψη της πρότασης Κομισιόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στις υπόλοιπες τροπολογίες. 5. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για να αλλάξουμε την 72 παρακαλώ. ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ και την 73. Πέρας. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά αποχές τη 49 παρακαλώ ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές και εδώ να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στους συζητητές. Φτάσαμε στο τέλος της ε, ψηφοφορίας και της πρωινής μας συνεδρίασης. Θα σας δούμε λοιπόν το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ που συνεργαστήκαμε τόσο καλά.